και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ε, συμβιβασμό, τον οποίο με ενθουσιασμό θα υπερψηφίσουμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας. Στρέφουμε λοιπόν αρχικά στους συντάκτες της προφορικής ερώτησης. Αλλά θα ήταν ε, καλό αν η Κομισιόν ήταν ήδη έτοιμη να ακούσει τους συντάκτες. Πρώτος λοιπόν στον κατάλογο, είναι πρώτη μάλλον, είναι η κυρία Χέραντς Γκαρσία για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που ήρθε και που έχει δείξει τόση μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές κρίσεις έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στην Ευρώπη εξαιτία του κόστους των πρώτων υλών, της ανισορροπίας που υπάρχει την συγκυρία που έχει περάσει τις τιμές των δημητριακών. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα όπως ε, και τα υπόλοιπα στην Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την ανακοίνωσή τη για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύη και να εκφράσουμε την ανησυχία μα για τόσα συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα. Και στην Ισπανία, τη χώρα μου, αλλά και σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για μια διαρθρωτική κρίση. Η αύξηση των τιμών των δημητριακών επιδίνωσε μια κατάσταση που ήδη είναι δύσκολη εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζεται. Τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι εγκαταλείπουν ε, τη γη οι αγρότες. Δεν θα έπρεπε όμως τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια όλο και θα μεγαλώνει η ζήτηση δεδομένου ότι βελτιώνεται το επίπεδο ζωής ε, των πολιτών. Στα πλαίσια λοιπόν της αναθεώρησης της ΚΑΠ τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προβλέπει για την κτηνοτροφία που είναι ειδικό τομέα. Μέτρα στην αγορά, αλλά και άλλα μέτρα τα οποία θα αποφύγουν μεταξύ άλλων τα μοντέλα εντατικής ε, κτηνοτροφίας πλήττονται ε, με το μελλοντικό καθεστώς ενισχύσεων. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν τον εφοδιασμό και θα φροντίσουν να είναι ο εφοδιασμός σε ζωοτροφές και θα βοηθήσουν να απελευθερωθούν τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν. Χαίρομαι πάντως που το σχέδιο αυτό ψηφίσματος αναφέρεται στο χείριο κρέας ιδιαίτερα και σε τομείς τα οποία δεν χαίρουν άμεσων ισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που μπορούν να επωφεληθούν από μέτρα στην αγορά για να ανακουφιστούν κάπως οι τομείς αυτοί. Ο κύριος Νίκολσον τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω το γεγονός ότι συζητείτε σήμερα αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Αυτή τη στιγμή ο τομέα τη κτηνοτροφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διανύει δυσκολίε που προκαλήθηκαν από διάφορου παράγοντε, αύξηση του κόστου παραγωγή, ανταγωνισμό αθέμητο από τρίτε χώρε και βέβαια διάφορα ζητήματα που συνέβαλαν στο αυξανόμενο κόστο των ζωοτροφών δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της ξηρασίας στην ε, Αυστραλία ή της κακοκαιρίας στην ε, Ρωσία. Όμως πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πιο επαρκείς όσον αφορά τις πρωτεϊνούχες ε, καλλιέργειες. Εξαρτώμεθα υπερβολικά από τρίτες χώρες για τις ζωοτροφές μας και πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες μας οι ίδιοι. Ωστόσο η κατάσταση που ισχύει είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε πολλές από τις ζωοτροφές μας και επανειλημμένως έχω πει ότι πιστεύω Πιστεύω πως η διαδικασία βελτίωσης νέου είδους ε, τροφών ε, γενετικά τροποποιημένων παίρνει πάρα πολύ καιρό. Επιγόντως πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Ένωση θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες τιμές, πτυτικότητα των τιμών και αβεβαιότητα για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Να αναφέρω σύντομα πώς ε, επηρεάζονται οι πτυνοτρόφοι, η πτυνοτροφία. Ε, εκείνοι πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση γιατί το κόστος αυξάνεται και η τιμή του κρέατος, ε, του, των πουλερικών αλλά και του χοιρινού ε, πέφτει διαρκώς. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί η κατάσταση. Η παραγωγή βόλου κρέατος εγωπροβάτων... Ε, Όλοι, όλοι χάνουν. Όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι χάνουν. Υποφέρει ολόκληρο ο τομέα αυτή τη στιγμή. Τέλος όμως πρέπει να πω όμως ότι ο καταναλωτής θα πληρώσει. Διότι τελικά άμα σταματήσουν να παράγουν κτηνοτρόφοι, τι θα κάνουμε. Θα χρειαστεί να εισάγουμε όλο αυτό το κρέας με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να έχουμε φτάρκια όσον αφορά την προμήθεια τροφίμων στην Ένωση. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό πραγματικά θα είναι εις βάρος μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αποδοτικότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής συνδέεται με το κόστος της οτροφής. Ε, δεδομένου ότι οι τιμές είναι ασταθείς όσον αφορά τις πρώτες ύλε, αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τις ζωοτροφές βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Ο κτηνοτροφικός τομέας περνάει δύσκολες στιγμές, κυρίως το χείριο κρέας. Η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών σημαίνει 60% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μέσα σε δύο μήνες αυξήθηκαν τα δημητριακά κατά 50% όσον αφορά τις τους. Δεν υπάρχει λοιπόν ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση για την παραγωγή, υπερβολική παραγωγή, αλλά από παράγοντες ξένους από εμά, με κερδοσκοπικά φαινόμενα να ακολουθούν και να κινδυνεύουν τα αποθέματά μας. Εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι βάζει από την παρέμβαση από θέματα δημητριακών στην αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ καλό. Ένας φόρος στην εξαγωγή δημητριακών, όπως είχαμε πει το 1994 και το είχαμε κάνει, θα ήταν μια λύση. Πάντως, η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν είναι δυνατόν να φτάνει ε, στα ράφια των μαγαζιών οι παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες χωρίς πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καταλαβαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα που ελπίζουμε ότι θα πάρει και θα τα συμπεριλάβει στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία, να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να ευνήσουμε τον ανταγωνισμό του κτηνοτροφικού τομέα και να φροντίσουμε να του δώσουμε την αξία που του πρέπει. Υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να ζητήσω να μπουν σε εφαρμογή και μέτρα όσον αφορά το χείρο κρέας. Επιστροφέ, για παράδειγμα. Η Επιτροπή λέει ότι δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο από την κατάσταση του τομέα. Όμω, του τελευταίου μήνε η τιμή του χειρίου κρέατος έχει μειωθεί και τα χρήματα που παίρνουν τελικά η παραγωγή χειρίου κρέατος είναι πάρα πολύ... Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί διαχειρισμού του, διαχείρισης ε, της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Σιόλος έχει τώρα το λόγο για να απαντήσει. Θα δώσω την απάντησή μου σε δύο τμήματα, γιατί όντως τα προβλήματα του τομέα της κτηνοτροφίας συνδέονται με την κατάσταση των τροφίμων, δηλαδή την κατάσταση της αγοράς δημητριακών. Θα αναφερθώ επίσης και στον μηχανισμό που έχουμε σκεφτεί για τον τομέα της κτηνοτροφίας τον ίδιο. Η Κομισιόν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στην αγορά δημητριακών και τις επιπτώσεις που αυτό έχει για την κτηνοτροφία. Ε, σημαντική αύξηση έχει διαπιστωθεί στη τιμή των δημητριακών λόγω της έλλειψης ε, ε, προμηθειών κυρίως στις χώρες της ε, Μαύρης Θάλασσας. Και έτσι είδαμε το κριθάρι και τη βρώμη να αυξάνονται μέχρι στα 200 ευρώ τον τόνο. Αυτή τη στιγμή το κόστος μένει κάτω από τις τιμές ρεκόρ που διαπιστώθηκαν το 2000, που σημειώθηκαν μάλλον το 2008. Η, η διαφορά στην συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο φυσικά θέτει ε, άλλο ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αγορά και το ευρώ. Παρά λοιπόν το έλλειμμα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, τα επίπεδα Εσοδεία είναι τα ίδια και ικανοποιητικά χάρη στη... έχουμε αποθεματικά δηλαδή χάρη στα δύο τελευταία χρόνια. Η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά μέσο όρο 276 εκατομμύρια τόνους και αν προσθέσουμε και τα αποθέματα έχουμε ένα πλεόνασμα 60 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με τις προβλέψεις ε, χρήσης. Τα στόκ παρέμβασης ε, ανέρχονται σε 5,6 εκατομμύρια ε, τόνους δημητριακών και βασικά είναι κρυθάρι. 8 εκατομμύρια τόνοι είναι είναι αυτά που έχουν μπει σε αποθεματικό και θα διανεμηθούν το 2011 υπέρ των λιγότερων προνομιούχων και ε, αν δεν χρησιμοποιηθούν θα χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική αγορά. Θα τοποθετηθούν στην αγορά ήδη από το τέλος αυτής, αυτού του μήνα. Και επίσης 100, μάλλον κάποια ε, άβληση της κατάστασης, κάποια μείωση της έντασης ε, παρατηρήθηκε μετά την ανακοίνωση αυτού του μέτρου από πλευράς της Κομισιόν. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ανησυχίες δεν, δεν δικαιολογούνται γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει πρόβλημα προμήθειας στην αγορά δημητριακών. Η υψηλή τιμή των δημητριακών δεν οφείλεται σε έλλειψη ε, παροχής στην αγορά. Στον τομέα λοιπόν της κτηνοτροφίας έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα του χείριου κρέατος και των πουλερικών. Τα περιθώρια εξαρτώνται πολύ από το κόστος των τροφίμων. Οι τιμές στον τομέα της πτηνοτροφίας είναι ανώτερες από τον μέσο όρο μακροπρόθεσμα και φαίνεται να αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους, την πτώση μάλλον του κόστους των τροφίμων. Εξάλλου ακολουθείται προς, με επιδοτική τάση η εποχιακή ε, πορεία, η εποχιακή τάση. Η παραγωγή λοιπόν απορροφάται καλά από την εσωτερική αγορά και από τις εξαγωγές. Ανάμεσα στον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2011 οι εξαγωγές χειρίου κρέατος αυξήθηκαν κατά 10% και οι εξαγωγές ε, πουλερικών κατά 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο της περασμένης χρονιάς. Είχαμε μια περίοδο δηλαδή που παρά το πρόβλημα των τιμών η παραγωγή παραγωγή χειρίου κρέατος και πουλερικών ε, μπόρεσαν να εξάγουν. Ωστόσο, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά και μόλις θα χρειαστεί απαραίτητο και σκόπιμο θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να παρέμβουμε στην αγορά διότι για τον τομέα της κτηνοτροφίας υπάρχουν δύο διαθέσιμα μέτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή είτε επιστροφές στις εξαγωγές είτε ε, η αποθήκευση. Τώρα, για τι επιστροφέ στι εξαγωγέ δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να είναι αποτελεσματικό αυτή τη στιγμή, γιατί η παγκόσμια τιμή είναι υψηλή. Άρα δεν δικαιολογείται να επιδοτούμε για τι εξαγωγέ. Το πρόγραμμα των εξαγωγών ε, μπορεί να χρειαστεί να παρέμβουμε, γιατί υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στο δολάριο και το ευρώ. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει μονάχα τον γεωργικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση, η ισοτιμία δηλαδή μεταξύ δολαρίου και ευρώ και με βάση αυτό Εάν έχουμε πλεονάσματα στην κοινοτική αγορά, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για μέτρα αποθήκευσης. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο πλεόνασμα κρέατος στις ευρωπαϊκές αγορές και γι' αυτό και το μέτρο της αποθήκευσης δεν ε, συζητείται. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε την δυνατότητα, την πιθανότητα χρήση αυτού του μέτρου. Όσον αφορά την πτυτικότητα, είναι ένα θέμα το οποίο ε, συζητείται για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ του 2013, όπου προβλέπεται να προτείνουμε μηχανισμού που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα το θέμα τη πτυτικότητα των εισοδημάτων των ε, γεωργών. Το θέμα τη διαφάνεια το μελετούμε αυτή τη στιγμή με τον Επίτροπο Ταγιάννη, τη διαφάνεια για την τροφική αλυσίδα, για να δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε διευκρινήσεις και έτσι να αποσαφινιστεί και η κατανομή της προστιθέμενης αξία. Αυτά μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή ως απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε και τώρα περνάμε στη συζήτηση. Να θυμίσω και πάλι στους συναδέλφους ότι πρέπει να παραμείνουν στο χρόνο ομιλία τους γιατί διαφορετικά θα πιεστούμε καθώς θα φτάνουμε στην ώρα των ψηφοφοριών. Πρώτον, λοιπόν, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων έχουμε τον κύριο Ντες για 1,5 λεπτό εξ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σημαντικό σημερινό ψήφισμα προσπαθεί να βοηθήσει τον, ε, την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και ε, χαιρετίζω την κυρία Χέρενς για αυτή την πρωτοβουλία διότι ο στόχος μας δεν είναι να καταστρέψουμε την Ευρώπη ή να καταλύσουμε την νομοθεσία αλλά να υπάρχουν δίκαιες ε, καταστάσεις στην αγορά κατά τρόπον ώστε ε, η διατροφή του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων στην Ευρώπη να μπορέσει να είναι εξασφαλισμένη. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη κάθε μέρα να προβαίνει σε νέα νομοθετήματα που καλύπτουν την τελευταία λεπτομέρεια και οι κτηνοτρόποι να πρέπει να ανταποκρίνονται, να λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα ασφάλειας ασφαλείας, ε, για το περιβάλλον, για το, ε, ε, το ζωικό κεφάλαιο και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους που υπερψήφισαν την πρόταση να πρέπει να σέβονται και οι εισαγωγές των ζωικών προϊόντων στην Ευρώπη τα ίδια μέτρα και σταθμάτα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες για τη διατύπωση αυτής της προφορικής ερωτήσεως και τη στηρίζουμε. Επόμενος ε, τώρα ο κύριος Ντεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητάμε αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν να θεσπίσει κατάλληλα αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που, αντιπροσω... που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας ε, της σήμερα στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι θα είναι γρήγορη η Επιτροπή για να μπορέσει να φτιάξει τέτοια μέτρα και ότι θα υπάρξουν και προτάσεις ώστε να περιοριστεί η πτυτικότητα των τιμών για ολόκληρο το γεωργικό τομέα. Ωστόσο, <clears throat> μπορούμε να διευκρινίσουμε περισσότερα πράγματα για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στου Ευρωπαίου κτηνοτρόφου. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν για το κτηνοτροφικό τομέα να ξαναδούμε την χρήση των ε, ζωικών αλεύρων για τα μη μυρικαστικά ζώα. Για, όπως ξέρετε, μετά από την κρίση της σπογκόδου εγκεφαλοπάθειας απαγορεύτηκε η χρήση αυτών των αλεύρων. Όμως σήμερα μπορούμε να πούμε μετά από τις μελετές που έχουν γίνει ότι μόνο για τα μυρικαστικά ζώα υπάρχει ο κίνδυνος, ενώ για τα υπόλοιπα όχι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργητικότητα σε αυτά τα ζώα και γι' αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα στην κατανάλωση αυτών των αλεύρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας αυτός είναι πολύ βασικός στην γεωργία γιατί οι κτηνοτρόφοι καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ένα βασικό ποσοστό ε, της υπαίθρου και η Ιρλανδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ε, βοήου κρέατος στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που εξαρτώνται από τις ζωοτροφές που βασίζονται στα δημητριακά και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, λάβει μέτρα για να αποφύγει ε, την αστάθεια των αγορών και θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ιδίως στις πιο μειονεκτικές περιοχές κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής των γεωργών, των κτηνοτρόφων, διαφορετικά θα μειωθεί και η παραγωγή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πλέον αυστηρή νομοθεσία σχετικά με ε, την ευημερία των ζώων και τα μέτρα ασφαλεία. Δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να μειονεκτούμε έναντι των ανταγωνιστών μας και θα πρέπει στον τομέα της κτηνοτροφίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν θα μειονεκτήσουν οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι και ότι θα μπορέσει να οδηγήσει την κτηνοτροφία της Ευρώπης σε ένα ευίωνο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ, ένα λεπτό για εν ονόματι των Πρασίνων. Κυρία Πρόεδρε ή κύριε Επίτροπε, όπως το 2007 οι τιμές των δημητριακών απογειώνονται και στο θέμα των κτηνοτρόφων βοήου κρέατος βλέπουμε να αυξάνονται πάρα πολύ τα έξοδά τους και να μειώνονται τα κέντρη του διότι βλέπουμε εδώ ότι ενώ ένα, μία μπριζόλα κάνει 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ο κτηνοτρόφος παίρνει 3 πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει και να απαγορεύσει την πώληση σε μία τιμή κάτω της τιμής κόστους για να μπορέσουν ε, να ε, διαμορφωθούν σωστά οι τιμές και οι κτηνοτρόφοι θέλουν ε, να ενισχυθούν οι οργανώσεις τους της αγοράς κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα θέματα και γι' αυτό ο Επίτροπος θα πρέπει να απαντήσει ή στα ερωτήματά μας διότι η Ευρώπη χρειάζεται Όλου όλους τους αγρότες της. Ευχαριστώ κύριος Σπογικόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, διότι ε, χαίρομαι ε, που αντιμετωπίζουμε την κατάσταση της κτηνοτροφίας η οποία είναι πολύ δυσμενής. Στο σημείο 15 του ψηφίσματος πιστεύω ότι όσον αφορά τις προδιαγραφές υγείας των ζώων θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να είναι υψηλότερες και τις υποστηρίζουμε αλλά η ευημερία των ζώων έχει σχέση με το κόστος και ε, το κόστος το αναλαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι πρέπει λοιπόν να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός διότι εισάγουμε ε, κτηνοτροφικά προϊόντα και κρέατα από τον τρίτο κόσμο χωρίς εκεί να σέβονται τις ίδιες προδιαγραφές διότι αν εισάγουμε εδώ προδιαγραφές θα πρέπει να απαιτήσουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά από στις τις χώρες οι οποίες θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους προς τη χώρα μας. Ο κύριος Λιαρίκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από τις τρέχουσες πολιτικές μας και να σταματήσουμε αυτή την πλήρη ελευθέρωση των αγροτικών αγορών που έχει σαν αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι, όπως είπαν πολλοί κι άλλοι, να κερδίζουν 700 με 800 ευρώ το μήνα, 700 με 800, ενώ οι τιμές στην κατανάλωση κρέατος θα αυξηθούν κατά 40%. Πρέπει να σταματήσουμε τις καταχρηστικές εισαγωγές και να σταματήσουμε να διαπραγματευόμαστε για αυτήν την ε, κακιά συμφωνία για την εισαγωγή 400.000 τόνων. Αντίθετα, πρέπει να έχετε το θάρρος να προστατεύσετε την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και να αποφασίζουμε εμείς και όχι η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου για την τύχη των κτηνοτροφικών μας ε, μονάδων. Χρειάζεται ρύθμιση, χρειάζεται να σταματήσει αυτός ο φωνικός ανταγωνισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέσετε τιμές βάσης σταθερές, δίνοντας περισσότερη αξία στην κτηνοτροφία που ε, γίνεται με ζώα τα οποία τρέφονται στα λιβάδια. Κύριε Επίτροπε, επίγει το θέμα. Δράματα εκτιλήσονται στην υπεθρό κάτι το οποίο κάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να χάνει την αξιοπιστία του. Ευχαριστούμε. Από το ΙΕΦΤ e ο κύριος Σκότα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι. Η πτυτικότητα των τιμών των δημητριακών έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τομέα των κτηνοτρόφων, τη κτηνοτροφίας αλλά και για του καταναλωτέ. Μιλάμε για πυρκαγιέ, για ξηρασία, για πλημμύρες, ε, καταστροφές οι οποίες μειώνουν την παραγωγή λόγω των ε, μεγάλων ε, βροχοπτώσεων αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον στην Ιταλία. Οι παραγωγοί δημητριακών που περιμένουν αύξηση των τιμών περιμένουν να δουν ποια θα είναι η παραγωγή τους και την αποθηκεύουν με συνέπεια την έλλειψη σε γεωργικά προϊόντα. Επίσης, μεγάλη αύξηση των τιμών των ε, δημητριακών ε, που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, πράγμα το οποίο οδήγησε και σε αύξηση της τιμής του κρέατος. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει γρήγορα μια παρέμβαση από την Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί η πτυτικότητα των γεωργικών προϊόντων μέσω των καινοτόμων μέτρων που προβλέπει η νέα ΚΑΠΗ. Είναι απαραίτητο να εμποδιστούν οι κερδοσκοπικές πρακτικές στον τομέα της γεωργίας για να εγγυηθούμε τα εισοδήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων και για να εγγυηθούμε και στους καταναλωτές υγιεινά προϊόντα σε δίκαιες τιμές. Σας ευχαριστώ, μη συνδεδεμένο μέλος, ε, η κυρία Ντότζ, για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να καλέσω το Σώμα να στηρίξει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ψήφισμα που έχουμε σήμερα ενώπιόν μα. Είναι προφανέ ε, για εμά που προερχόμαστε από αγροτικέ περιφέρειες και που εδρεύουμε στην Γεωργική Επιτροπή ότι η κατάσταση πολλών κτηνοτρόφων αυτή τη στιγμή είναι βάσταχτη. Δεν είναι μια απόπειρα να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, ω συνέπεια θα αντιμετωπίσουμε ψηλότερε τιμέ στα τρόφιμα και θα εξαρτώμαστε περισσότερο από εισαγωγέ από τρίτες χώρε. Χώρε όπω η Κίνα ή η ΕΠΑ όλο ένα περισσότερο να γνωρίζουν την τη σημασία τη ασφάλεια στην ε, προμήθεια τροφίμων και γι' αυτό και αυξάνουν τη στήριξη που δίνουν στην γεωργία του. Στη Βόρεια Ιρλανδία η τιμή του βόλου κρέατος είναι πολύ πάνω από την... Ε, το κόστο παραγωγή. και όσο αυξάνεται η τιμή καθώ και οι επιπλέον απαιτήσει αυξάνονται τότε οι κτηνοτρόφοι ξεφεύγουν από την εκτινοτροφία, εγκαταλείπουν τα στις περιοχές, εγκαταλείπουν ε, τα ζώα και έτσι θα δημιουργηθεί έλλειψη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σημασία της ασφάλειας στα τρόφιμα και την αξία που έχουν οι κοινοτρόφοι και οι γεωργοί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, τα εμπόδια από τη Μερκοσούρ ε, έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Ε, ο τομέας της, της κτηνοτροφίας έχει επιβαρυνθεί μέσω της μεγαλύτερης αβεβαιότητας που τονίστηκε με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ. Μέχρι στιγμής οι παραγωγοί στην Βόρεια Ιρλανδία πιστεύουν πως τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι μόνο αρνητικά για τους Ευρωπαίους ε, γεωργούς και για την ποιότητα των τροφίμων που προσφέρουν Στου στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Τώρα ξεκινούν οι μεμονωμένοι ε, <coughs> ομιλητές και πρώτα ο κύριος Νικουλέσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, δεν είναι η γεωργία αλλά οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ουσιαστικά τα θύματα αυτής της κρίσης διότι ξέρουμε ότι η τιμή ε, των δημητριακών επηρεάζει την τιμή των Ζωτροφών και άρα το κόστος παραγωγής. Ε, μία αναλογική αύξηση των τιμών δεν είναι είναι δυνατή και οι ε, κτηνοτρόφοι δεν ε, έχουν τη σωστή τιμή. Ε, τα σπασμένα τα πληρώνουν δηλαδή οι καταναλωτές και θα πρέπει να επέμβουμε και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την διανομή. Αλλά υπάρχει γενική κρίση τώρα, μία μείωση της αγοραστικής δυνάμεως η οποία επηρεάζει και τον τομέα της κτηνοτροφίας και θα είναι δύσκολο για τους κτηνοτρόφους να εξασφαλίσουν ζωοτροφές το χειμώνα πράγμα το οποίο ε, θα παρατείνει την κρίση για να υπάρχουν οι αναγκαίες κτηνοτροφές και σωστές τιμές θα πρέπει να ανεβάσουμε την τιμή παρέμβασης και συμφωνώ με τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να υπάρχουν ε, γενετικά ε, τροποποιημένοι οργανισμοί για να εξασφαλίσουμε την αναγκαία διατροφή κατά τον χειμώνα και αυτή τη στιγμή θα πρέπει συγχρόνως να αναθεωρήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική η οποία πρέπει να είναι καλά χρωμοδοτημένη, ε, εξυγχρονισμένη για να μπορέσει να στηρίξει την αγορά. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι συνειδητοποιούμε τις τεράστιες δυσκολίες που διανύει ο τομέας της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη, κυρίως η χειροτροφία. Ε, γνωρίζουμε τόσα προβλήματα συμπεριλαμβάνοντας το ψήφισμα το οποίο αυτό ε, που συζητάμε και διαπιστώνεται ψηλό κόστος των δημητριακών. Αυτό είναι το ξεχωριστό στοιχείο. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε αυτή την κατάσταση. Είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε άμεσα χρησιμοποιώντα διαθέσιμους μηχανισμούς και γι' αυτό το θέμα ε, χαιρετίζω την απόφαση της Κομισιόν να βάλει στην αγορά 2,8 εκατομμύρια τόνους που είναι σημαντική κίνηση αλλά όχι επαρκή. Θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα μέσω και, μακρο... και βράχη πρόθεσμα για να αντιμετωπίσουμε το κόστος ε, των δημητριακών. Μάλιστα ο κύριος Επίτροπο επεκστίασε εκεί το πρόβλημα και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα κάπου που τώρα θα, θα ξεκινήσει. Λαμβάνοντας υπόψη τις ε, συστάσεις που εμείς ε, σας κάνουμε στο ψήφισμα που συνυπογράφουν διάφορες ε, πολιτικές ομάδες θα πρέπει να τις λάβετε υπόψη γιατί είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, Επίτροπε. Χόσλινγκ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλά εδώ προτείνονται πρότυπα με τα οποία δεν συμφωνούμε ε, ε, όταν διευκολύνουμε τις εισαγωγές ε, ε, δεν ε, λύνουμε την κρίση στην κτηνοτροφία πρέπει να βελτιώσουμε την, παραγωγή πρωτεϊνών και θα πρέπει ορισμένα πράγματα να αλλάξουν και δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι αμφισβητούν τον συμβιβασμό στον οποίο συμφώνησαν όλες οι πολιτικές ομάδες και ε, ε, προσπαθούν να αλλάξουν τα θέματα των εισαγωγών διότι βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πλήττονται περισσότερο από την κρίση και υπάρχει μια κατάσταση στην κτηνοτροφία η οποία δεν είναι σωστή η οποία δεν είναι δίκαιη για τους κτηνοτρόφους και επιπλέον βλέπουμε έχουμε 450 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν στο ίτερ και θα ήθελα να μου πει ο Επίτροπος γιατί γίνεται αυτό. Η κυρία Ντεμπρίν για ένα λεπτό. η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών του, ε, ε, ε, του σιταριού και του κρυθαριού επηρεάζουν την ε, κατάσταση η οποία είναι ήδη κακή στον τομέα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και επιτείνουν την αύξηση των τιμών. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει πολιτικές για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την τιμή των ζωοτροφών και των ε, ε, κτηνοτροφικών προϊόντων. Και αντιλαμβάνομαι ότι ε, για το 2012-2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα νέο μέτρο, αλλά τώρα χρειαζόμαστε τα μέτρα αυτά. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σε, Συμφωνώ και θεωρώ ότι η παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική διότι αυτή τη στιγμή ε, δεν αντιμετωπίζεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχει μία ε, στην χώρα μας ένα σύστημα αναγνωρίσεως των προβάτων πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε όλες τις χώρες και υπάρχει υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός οπότε ε, θα πρέπει ε, να υπάρξει μια τροπολογία η οποία να καλύψει την επιστροφή των χρημάτων τα οποία ξοδέψαμε για αυτό το άδικο μέτρο το οποίο δεν σεβόνται άλλες χώρες. Σχετικά με τις ε, συμφωνίες με τις χώρες του Μερκοσούρ δεν είμαστε ευτυχείς σχετικά με αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. ένα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μία κρίση στο χώρο και υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κρίση αυτή. Ορισμένοι λέγουν ότι ένας από τους λόγους είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός και επιπλέον ο κίνδυνος των εμπορικών συναλλαγών με το Μερκοσούρ. Αλλά άλλοι μιλούν για τη γρήγορη αύξηση των τιμών των σιτηρών. Ήταν κάτι που είχαμε προβλέψει. Το είχαμε θίξει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κινήθηκε. Έχουμε λοιπόν μία επιστροφή Τη της ε, παρεμβάσεως, διότι θα πρέπει η εμπορία των σιτηρών να μην είναι μόνο αντικείμενο της Ευρώπης αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της ε, κερδοσκοπίας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους καταναλωτές. Το κόστος όλων αυτών των μέτρων το πληρώνει ο Ευρωπαίος καταναλωτής το 2003 έως 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση πούλησε αποθέματα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ήταν ε, τότε ε, η τιμή των στυρών πολύ χαμηλή. Εάν είχε αγοράσει όμως η Ευρώπη τότε σιτηρά θα μπορούσε τώρα να τα χρησιμοποιήσει. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα κέρδη αλλά πρέπει να δούμε και τις ανάγκες ανάγκες των χωρών σαν το Πακιστάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ε, πρωτοβουλία του ε, Επιτρόπου Τσόλος σύμφωνο ότι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την αστάθεια των τιμών στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό παρεμβάσεως και προστασίας. Επίσης οι τιμές των σιτηρών ανεβαίνουν και δεν υπάρχουν αρκετές πρωτεΐνες στην Ευρώπη. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στον τύπο. Υπάρχει και ένα διαφορετικό θέμα ε, στην ε, κρίση αυτή. Δηλαδή υπάρχουν στρεβλωμένοι μηχανισμοί ε, προστασίας και η παραγωγή δημητριακών έχουν μεγαλύτερα κέρδη από ότι οι κτηνοτρόφοι οι δεν, ε, δεν τα βγάζουν πέρα διότι έχουν υποχρεωθεί να αναλάβουν μεγάλες, ένα μεγάλο ποσοστό των αυξήσεων των τιμών. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσόλος, κυρίες και κύριοι όσον αφορά τον, ε, ε, τη συνάδελφο Γκαρσία θα ήθελα να την ευχαριστήσω και θα ήθελα να αναφερθώ εις ε, την κατάσταση της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές γιατί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχει κοινοτροφία όπου δεν μπορούν πλέον να εξασκήσουν συνεχίσουν το επάγγελμά τους διότι αν δεν υπάρχουν ζωοτροφές ε, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη ποικιλομορφία και εδώ αναφέρομαι και στη γαλακτοκομία και άλλωστε και στη γαλακτοκομία σε ορεινές περιοχές όπου ε, θα πρέπει να επέμβουμε και γι' αυτό στην γεωργική πολιτική πρέπει να προσέξουμε διάφορα πράγματα. Καταρχήν θα πρέπει να συνδυαστούν οι ε, ενισχύσεις με την παραμονή στις ορεινές περιοχές, δηλαδή ε, θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να στηριχτούν και να υπάρχει μια ποιοτική πολιτική η οποία θα βασιστεί ε, σε προϊόντα ε, τα οποία θα είναι υψηλού επίπεδου ε, για να μπορούν και οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών να έχουν μια πρόσβαση στην αγορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιθανότατα προχωρούμε προ μια νέα φούσκα στα αγορέ των αγαθών. Οι τιμέ στι διεθνεί αγορέ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 16% από τον Ιούνιο. Οπότε δεν έγιναν τόσε συναλλαγέ στι αγορέ των futures, ούτε ε, κυκλοφορούσαν τόσα πολλά χρηματοπιστωτικά ε, μέσα. Οι πολύ τα χαμηλά επιτόκια οδηγούν και ψάχνουν, ε, θέτουν χρήμα στην αγορά αγορά, το οποίο αναζητά επενδύσεις χωρίς όμως πραγματικό αντίκτυπο στην ε, πραγματική οικονομία. Έχουμε ε, σπάσει ρεκόρ στις διαπραγματεύσεις αγορών στη Σόγια, στον Αραβόστο και στο Σιτάρ. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η μεταφορά αυτών ε, στις τιμές της πραγματικής αγοράς, χωρίς όμως να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά σε δημητριακά. Είμαστε ήδη σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τις εξαγωγές του, του αγροκοινοτροφικού τομέα που πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ξανασηκώσει κεφάλι. Γι' αυτό και ακριβώς πρέπει να τεθεί τέλος στην, στην κερδοσκοπία για τα τρόφιμά μας. Και γι' αυτό και ρωτώ τι θα κάνει η Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Νταντάν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι κόσμο είναι αυτό ο κόσμο τη Γεωργίας. Πριν από ένα χρόνο, εδώ σε αυτό το ημικύκλιο, Όλοι μιλούσαμε για το σύνολο της παραγωγής. Σήμερα έχουμε έναν τομέα, τα δημητριακά, που πάνε καλύτερα από τους άλλους. Μπράβο για τα δημητριακά. Όμως από την άλλη υπάρχουν συνέπειες τραγικές σε έναν άλλο τομέα που είναι η κτηνοτροφία. Το πραγματικό ερώτημα σήμερα είναι ότι ο αγροτικός κόσμος δεν καταφέρνει να μεταφέρει προς τον καταναλωτή τα δικά του βάρη. Γι' αυτό πρέπει, όπως το είπαμε και σήμερα το πρωί, να ευνοήσουμε την οργάνωση των παραγωγών έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο βάρος απέναντι στους πελάτες τους και απέναντι στη μεγάλη διανομή. Όμως, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά, δεν βοηθάει. Πώς να εξηγήσουμε ότι για δεκαετίες και για χρόνια λέμε ότι η Νότια Αμερική βαραίνει στην παραγωγή και κατεβάζει τις τιμές. Και σήμερα στις χώρες αυτές που η τιμή αυξάνει, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο και για τους δικούς μας παραγωγούς. Φυσικά και τα βάρη αυξήθηκαν, αλλά η, παρα... η τιμή στην παραγωγή δεν αυξήθηκε. Πώς να αποσιοποιήσουμε επίσης όλα αυτά, όλες αυτές τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες, στις χώρες μας. Φταίνε τα κράτη σε βαθμό. Αλλά το dumping αυτό συμμετέχει στην αποσταθεροποίηση των αγορών. Γι' αυτό και η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Ναι, πρέπει να βρει λύσει. Οι παραγωγοί δημητριακών το γνωρίζουν, καταλαβαίνουν ποια είναι η κατάσταση που πλήττει τους κύριους πελάτες τους που είναι οι κτηνοτρόφοι και είναι διατεθειμένοι να φροντίσουν να υπάρξει μια συμφωνία. Εσείς κύριε Πίτροπε θα στηρίξετε μια τέτοια συμφωνία. Ο κύριος Κέλλη τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επιτροπή, για άλλη μια φορά εδώ συζητάμε για τους αγρότες και για την καταστροφή των αγορών, για τις δυσλειτουργίες που επικρατούν στις αγορές μας, για το χείριο κρέας ιδιαίτερα. Θέλουμε ένα δυνατό σύστημα των αγορών και ελπίζουμε ότι ο Επίτροπος θα φροντίσει να ακούσει την έκκληση των πολιτικών μονάδων που γίνονται εδώ στα πλαίσια της νέας περίοδου μέχρι το 2013. Οι ρυθμίσεις έχουν, ε, πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνει πιο ανταγωνιστικό ο τομέας και όχι το αντίθετο. Με ένα σύστημα υπέρ του περιβάλλοντος που εφαρμόζεται και για τις αγωγές μας από τρίτες χώρες. Το ότι δεν υπάρχει αυτάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι σοβαρό όχι μόνο για το Βόλιο κρέας αλλά και για τα πουλερικά και για το χείριο κρέας. Εξαρτάται από το πόσο σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε εμείς την κατάσταση αυτή. Ω Κοινοβούλιο πρέπει να παρεμβαίνουμε κάθε φορά που βλέπουμε ότι επήγει το ζήτημα. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο αν φροντίσει για την παρέμβαση, για αποθέματα την παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς, βόηο, χείριο και πουλερικά. Ευχαριστώ τελείωσε το τμήμα αυτό της συζήτησης. Μας έχουν ζητηθεί πάρα πολύ να πάρουν το λόγο στη διαδικασία του Catch the όμως επειδή πιέζει ο χρόνος μόνο πέντε ομιλητές θα επιτρέψω, φροντίζοντας να τηρήσω μια πολιτική ισορροπία. Να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ για να μπορέσουμε μετά να ακούσουμε και την απάντηση του Επιτρόπου. Πρώτος στον κατάλογό μου είναι ο κύριος Καλανάφσκι. Πρόεδρε, Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Τα όσα συνέβησαν φέτος είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ότι δηλαδή χρειάζεται να έχουμε πάντα τα απαραίτητα αποθέματα σε δημητριακά για τη προσκάρτη τη σταθερότητα τη αγορά. Αυτά αφορούν πολιτικέ αποφάσει που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ε, χρειαζόμαστε διαφορετικέ πηγέ πρωτεϊνών για να πρωτεϊνούχων ε, προϊόντων για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να τονώσουμε την αγορά και την παραγωγή μας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί μας, οι κτηνοτρόφοι, θα έχουν πρόσβαση σε ζωοτροφές. Γι' αυτό και στηρίζω την ιδέα της δημιουργίας ενός μίνιμουμ κατοφλίου σόγιας ε, γενετικά τροποποιημένη. Ο Δύο είναι, δύο είναι οι απειλές αυτή τη στιγμή για την ε, παγκόσμια κτηνοτροφία και διατροφή. Από τη μία έχουμε τα μονοπόλια των σπόρων που έχουμε δει τα μεταλλαγμένα και τις επιπτώσεις του στην Ινδία, τις καταστροφικές επιπτώσεις. Από την άλλη έχουμε τα παιχνίδια των κτηματοπιστωτικών οργανισμών ε, με τις τιμές των βασικών προϊόντων. Το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγή σιτηρών. Το 2008, παράλογα, αν δεν το εξηγήσουμε λόγω των χρηματοπιστωτικών παιχνιδιών, είχαμε και τη μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Επιστητική κρίση που οδήγησε σε κοινωνική αναταραχή και στην απώλεια της ζωής πολλών συνανθρώπων μας. Θα πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα δύο θέματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους τοπικούς πόρους να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στους πόρους για τους καλλιεργητές, να έχουμε χαμηλότερες τιμές και για τους κτηνοτρόφους. Και θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη λειτουργία των κτηματοπιστωτικών οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέει η κυρία Μπαράντικα, Πρέπει να έχουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές. Άλλοι αυξάνουν τις τιμές, κάτι από το οποίο πλήττονται άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την επαρκή χρηματοδότηση μετά το 2003 για να έχουμε βιωσιμότητα των ε, αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα επίσης για τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν ε, μέτρα βιώσιμα. Έχουν μια παραγωγή που βασίζεται σε βιώσιμους τρόπους παραγωγής. Έπειτα να ευνοήσουμε τις μειονεκτικές περιοχές. Τέταρτον, να φροντίσουμε οι εξαγωγέ που μα έρχονται από τρίτε χώρε να τηρούν τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ για να μην υπάρχει αθέματο ανταγωνισμό. Τέλο, ζητάω από την Επιτροπή να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αγροτών σε όλε τι εμπορικέ διαπραγματεύσει για να μην τίθεται σε κίνδυνο ο δικό μα κτηνοτροφικό τομέα. Αλλιώ, η Ευρώπη θα είναι ένα χώρο χωρί γεωργία και χωρί κτηνοτροφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στίβενσον τώρα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει πλήξει πολύ τους ε, σκοτσέζους κτηνοτρόφους και θα πρέπει να μειώσουμε το ρυθμιστικό ε, βάρος διότι δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε μεγαλύτερη γραφειοκρατία για τους κτηνοτρόφους από ότι έχουμε για τους εισαγωγείς και εφόσον εισάγουμε ε, πάρα πολλά ε, ε, ε, πάρα πολλά προϊόντα από το εξωτερικό χωρίς να σεβόμαστε ε, τις ίδιες προδιαγραφές. Αυτή τη στιγμή το κόστος του βρετανικού βοήου κρέατος είναι κάτω από την τιμή παραγωγής, χάνουν οι κτηνοτρόφοι μας μεγάλα ποσά και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την διολύστηση. Ευχαριστώ. Κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η αύξηση των τιμών των Δημητριακών είναι γεγονό το οποίο επιδεινώνει την κρίση στον τομέα τη συνοτροφία. Η ΚΑΠ και οι εμπορικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφαλίζουν δίκαια εισοδήματα στου ε, ε, γεωργού, ούτε αποφεύγουν. Αντίθετα, επιδεινώνουν το κόστο ε, τη παραγωγή και την πτυτικότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Αυτή η πτυτικότητα έχει, οφείλεται σε κάποιου λόγου που δεν είναι φυσιολογικοί ο πρώτος και καλύτερος λόγος είναι η κερδοσκοπία. Ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Ε, θα είναι περιορισμένα εάν δεν περάσουμε από την απαγόρευση των ε, παραγωγών χρηματοπιστωτικών προϊόντων ε, που οδηγούν στην κερδοσκοπία, που επιτρέπουν μάλλον την κερδοσκοπία. Η ασφάλεια σε τα τρόφιμα απαιτούν παραγωγή ε, δική μας ε, τροφίμων και παροχή τους στην αγορά. Απαιτούν μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά, χωρίς τους οποίους η, παρέμβα... η πτυτικότητα των τιμών θα συνεχίζεται. Ε, μόλις ένα, ένα μικρό νούμερο μεγάλων παραγωγών θα επιβιώσουν από αυτή την κατάσταση. Τέλος, ο Επίτροπος Σιόλος. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, με τα μεγάλη χαρά βλέπω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για έναν τομέα που είναι ουσιαστικός όχι μόνο για την προστασία της αγοράς αλλά για την ισορροπία των περιοχών μας και πρόκειται για την κτηνοτροφία. Πολλά από τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία εφήγησαν θα απαντηθούν μέσω των προτάσεων που θα κάνει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής και είναι προτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε και στο Κοινοβούλιο συντομότατα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Τότε θα συζητήσουμε και το θέμα της δικαιοσύνης των επιπέδων στηρίξεων στους διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και της ε, κτηνοτροφίας και ιδίως σε δύσκολες και μειονεκτικές περιοχές. Θα συζητήσουμε και τον μηχανικό για τη διαχείριση της ασταθίας των εισοδημάτων. Βεβαίως υπήρξαν ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν και θα ήθελα να απαντήσω. Το πρόβλημα των τιμών δημητριακών και των αποθεμάτων επεμβάσεως, πράγματα οποία είχαμε στο παρελθόν, όχι όμως τώρα γιατί οι τιμές είναι πιο υψηλές. Μία επέμβαση στην αγορά δεν αιτιολογείται εάν η τιμή είναι υψηλή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε να βρούμε άλλους μηχανισμούς και αν ε, ε, ε, κάνουμε αποθέματα δεν θα είναι τα αποθέματα επεμβάσεως ε, που θα ε, χρησιμοποιούνται στην αγορά και να ε, ασχοληθούμε με ένα πεδίο πιο ευρύ πέραν της Ευρώπης διότι και τώρα έχει μεγαλώσει ο χώρος αυτός. Όσο για το ίτερ κύριε Χόισλινγκ δεν σημαίνει ότι επειδή το 2010 δεν χρησιμοποιήθηκε ένα ποσοστό του προπολογισμού της Γεωργίας και θα χρηματοδοτήσει το ίτερ ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε τη Γεωργία διότι ε, τα χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο ίτερ είναι, χρήσιμα, είναι χρήματα τα οποία έμειναν αχρησιμοποιητά διότι δεν χρειάστηκε. Έχουμε όμως επαρκή, επαρκή πόρους για να αναλάβουμε τα μέτρα τα οποία χρειαζόμαστε. Τέλος θα ήθελα να πω ότι το θέμα της ε, ασταθίας και ε, της επιρροής των των ε, τιμών ε, στην αστάθεια ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως και τα παράγωγα, χρηματοοικονομικά παράγωγα στη συνεργασία με τον συνάδελφο Μπανιέ και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία πρώτη συνάντηση της ομάδας υψηλού επίπεδου στο το θέμα αυτό που έχουμε οργανώσει από κοινού με τον Επίτροπο Ταγιάννη. Ευχαριστώ και τα υπόλοιπα θα συζητηθούν όταν θα συζητήσουμε την πρόταση αναθεώρησης της κοινή γεωργικής πολιτικής που θα κάνει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ολοκληρώσατε τη συζήτηση. Τέλος τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει σε λίγο. Λίγα λεπτά διάλειμμα. Παρακαλώ, καθίστε. Η Προεδρία θα κάνει μία ανακοίνωση